η, ομάδα του ΕΛΚ, οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλιστές μου έχουν υποβάλει αιτήσει για διορισμούς στις αντιπροσωπείες και τις επιτροπές. Εάν δεν λάβουμε σχόλια πριν την, απόφαση, πριν την έγκριση των πρακτικών, αυτοί οι διορισμοί θα γίνουν δεκτοί. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο από τις 9 μέχρι τις 1